Uh, λοιπόν, καλώς ήρθατε στην συνεδρίασή μας για να ψηφίσουμε και μόνο να ψηφίσουμε. Έχετε τις κάρτες για να ψηφίσετε, ελπίζω όλοι. Και αρχίζουμε αμέσως με την τροπολογία 15. Υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Τροπολογία 295 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά τη 295. Τη ψηφίζουμε την τροπολογία 295 ηλεκτρονικά. υπέρ ή κατά με το μηχάνημα. Πέρας. Απερίφθη με διαφορά τριών ψήφων. Τροπολογία 16 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Η 2.96 καταπίπτει. Συμβιβαστική G υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 301 καταπίπτει, πάμε στην 302 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τρο... Συ... Συμβιβαστική H υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική N υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 309 υπέρ κατά αποχές εγώ θα έλεγα ότι απορρίπτεται αλλά θα το ελέγξουμε ψηφίζουμε την 309 άρχεται η ψηφοφορία για την 309 πέρας και απερίφθη 310 υπέρ κατά Αποχές απορρίπτεται. 311 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται θα έλεγα εγώ έλεγχος ψηφίζουμε 311 και τώρα άρχεται η ψηφοφορία πέρας πέρας απεριφθεί 23 υπέρ 23 κατά Προχωρούμε 313 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 314 έχει αποσύρθει. Και η 315 επίσης. Πάμε τώρα στο κείμενο της Κομισιόν. Το άρθρο 2.1 υπέρ. Κατά αποχές δεκτό. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Α, να ψηφίσουμε. Είμαστε στην 22 και θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. με 26 ψήφους δεκτή. Πάμε στην 23 μαζί με την 321 υπέρ. Κατά αποχές δεν βλέπω. Πρέπει να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την 23 μαζί με την 321. Και άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας και απορρίπτεται με 26 ψήφους. Προχωρούμε 24 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Θα έλεγα, αλλά θα ελέγξουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 24. Άρχεται πέρας της ψηφοφορίας. Απερίφθη με έξι ψήφους διαφορά. Ή 25. Ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Αποχές. Μ, απορρίπτεται. Α, θα ελέγξουμε. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά την 25. Άρχεται η ψηφοφορία. Τροπολογία 25. Πέρας. δεκτή με διαφορά τεσσάρων ψήφων 322 υπέρ κατά αποχές δεκτή 324 υπέρ κατά αποχές δεκτή 320 όχι συμβιβαστική αι συμβιβαστική αι υπέρ κατά αποχές δεκτή 342 υπέρ κατά αποχές δεκτή Όχι. Η 342 κατέπεσε. Λόγω της ψήφισης της 309. Όχι. Ναι. Τέλο πάντων, σε συνάρτηση με το 309, ε, καταπίπτει 342, 26 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 343 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 27 υπέρ Α, όχι, όχι, δεν μπαίνει σε ψηφοφορία 27. Δεν θα την ψηφίσουμε. Ε, ε, α, όχι, θα μπει. Ψηφίζουμε 27. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Τροπολογία 344 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Η 345 καταπίπτει, η 346 καταπίπτει. Πάμε στην 28 και την 347 από κοινού. Όχι, καταπίπτει. Όχι, καταπίπτει. Πάμε στη συμβιβαστική J, υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Η K, συμβιβαστική υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 354 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 355 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 350 6 καταπίπτει. Πάμε στη συμβαστική L υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 360 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Η 361 καταπίπτει. 340 και 341 ταυτόσιμες τροπολογίες υπέρ. Κατά αποχές δεκτές. Συμβιβαστική M, υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 367, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Ή 30, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 31, υπέρ, κατά αποχές δεκτή 32 υπέρ κατά αποχές ε, θα έλεγα ότι ε, εγκρίνεται αλλά θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά την τροπολογία 32 άρχεται η ψηφοφορία πέρα της ψηφοφορίας και απερίφθη η τροπολογία 368 θα την ψηφίσουμε αυτή. Την ψηφίζουμε 368 υπέρ. Κατά αποχές θα έλεγα ότι είναι δεκτή. Πάμε στην 23 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική όμικρον υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 35 υπέρ κατά αποχές δεκτή 371 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται έλεγχος ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 371 άρχεται η ψηφοφορία και πέρας της ψηφοφορίας. Απερίφθη. Τρακόσα εβδομήντα. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 372. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 36 υπέρ κατά αποχές δεκτή 373 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 374 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική π υπέρ κατά αποχές δεκτή 38 υπέρ κατά αποχές δεκτή 376 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική Q υπέρ κατά αποχές δεκτή 40 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Α, θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά τη 40. Πέρας. Απερίφθη με διαφορά τριών ψήφων. Συμβιβαστική R. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 385 υπέρ κατά Αποχές. Απορρίπτεται. Α, έλεγχος. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά την 385. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Α, δεκτή. Συμβιβαστική S υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ε, συγγνώμη. Δεκτή, δεκτή, δεκτή. Συμβιβαστική τι υπέρ κατά αποχές δεκτή. 397 μαζί με την 398, 399 και την 400 έτσι υπέρ των τεσσάρων Είναι τέσσερις ταυτόσιμες τροπολογίες εδώ. Υπέρ λοιπόν, κατά αποχές δεκτές, 402, 403, 404, 402, 403, 404 υπέρ. Έχει καταπέσει 401. 402, 3 και 4. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτές. 41 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Α, έλεγχος στη 41. Άρχεται η ψηφοφορία, πέραση της ψηφοφορίας, 41, απερίφθη. 405 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 406 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 407 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Α, έλεγχος. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά τη 42. Και πέρασε της ψηφοφορίας επί τη 42 και έχει γίνει δεκτή με διαφορά μιας ψήφου. Συμβαστική γιου υπέρ κατά αποχές δεκτή. ή 411 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 412 υπέρ κατά αποχές δεκτή 413 καταπίπτει συμβιβαστική β υπέρ κατά αποχές δεκτή 418 μαζί με την 419 υπέρ κατά αποχές δεκτές 420 μαζί με την 421 υπέρ κατά αποχές δεκτές συμβιβαστική W υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβιβαστική X υπέρ κατά αποχές δεκτή 428 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται έλεγχος ψηφίζουμε την 428 άρχεται η ψηφοφορία πέρας και απερίφθη 429 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 430 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Α, έλεγχος ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την τεροπολογία 43 άρχεται η ψηφοφορία πέρας της ψηφοφορίας ε, ε, είναι μία παραπάνω στο έλεγχο, μία ψήφος παραπάνω. Ας δούμε τα αποτελέσματα. Λοιπόν, με δύο ψήφου διαφορά καταρρύπτεται και πάμε συμβαστική Y υπέρ κατά αποχέ δεκτή ή 45 υπέρ κατά αποχέ. απο, όχι, αποχές θα έλεγα δεκτή Έλεγχο. ψηφίζουμε ηλεκτρονικά τη 45 άρχεται η ψηφοφορία πέρας τη ψηφοφορία και απορρίπτεται. 434 υπέρ κατά αποχές θα έλεγα ότι απορρίπτεται. Προχωρούμε στη συμβαστική ΑΑ υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική ΑΒ υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ε, συμβαστική ΑΣΥ, AC, ε υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Συμβιβαστική AD, ε υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Συμβιβαστική AE, αε, υπέρ κατά αποχές δεκτή. Λοιπόν, δεν την ψηφίζουμε την 58, ούτε την 458, ψηφίζουμε την 59 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή, συμβαστική ΑΕΦ υπέρ κατά αποχές δεκτή. Και ε, τροπολογία 70 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική AG υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική AH υπέρ κατά αποχές δεκτή. Η 87 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 88 κατά πίπτη, Πάμε στη συμβαστική AI. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 98 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 328 και 329 μαζί υπέρ, 98 εγκρίθηκε. Άρα πάμε στα 328 και 329 μαζί. Καλώς ψηφίζουμε. 328 και 329 μαζί υπέρ. Κατά. Α, αποχές εγκρίνονται. Εγκρίνονται μάλλον. 330 και 331 μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 332 και 333 μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, απορρίπτονται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τα 332 και 333. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. εγκρίνονται 335 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 334 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται έλεγχος για το 334 από το δεν σηκώνετε τα χέρια σας. Έλεγχος για το 334. Ψηφίζουμε το 334. Πέρασε. Εγκρίνεται. 338 και 339 μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 99 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Συμβαστική α κάπα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παναβάρτος α κάπα ε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 116 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική AL υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 127 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική AN υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ΑΕΝ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. AO υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 139 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική AP υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 499 πρέπει να την ψηφίσουμε. Ναι, πρέπει να ψηφίσουν την 499 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος για την 499. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται 32-16 συμβαστική A Q. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 150 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική A R υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική AS υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική AT υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και πάμε στο 162 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. AU συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική A Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 175. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. AV. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 191 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική A 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 510 καταπίπτει. Και η 511 Λοιπόν, στη συμβαστική AY υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 522 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Okay, we vote on amendment 337. Those in... 337 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 337 καταπίπτη και πάμε στην συμβαστική AZ υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική BA υπέρ. Κατά Αποχές. Εγκρίνεται. Z συμβαστική υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 553. υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 554 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτωται. 555 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 555 έλεγχος ψηφίζουμε πέρας Και εγκρίνεται με τρει ψήφου διαφορά και πάμε τώρα 231 πέρα. Κατά αποχές απορρίπτεται 232 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 233 υπέρ. Έλεγχος για το 232. Ψηφίζουμε. Εγκρίνεται. 233 υπέρ. Κατά αποχές. Έλεγχος. Ψηφίζουμε. Πέρασα. Απορρίπτεται. Ένα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική α. Ε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 239 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται έλεγχος για το 239 ψηφίζουμε and it is rejected. Πέρασε, απορρίπτεται. Uh, we are on uh, amendment 3, those in favor. 3, υπέρ, κατά, αποχές Απορρίπτεται. 240 those in favor. 240 υπέρ. Against, abstentions carried, 241. Εγκρίνεται, είπαμε 240. Α, θέλετε 240 έλεγχο. Μάλιστα. Επαλήθευση. Για το 240. And the vote is now closed. And it's rejected. Ε, Απορρίπτεται 241 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 242 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 243 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται έλεγχος για το 243 ψηφίζουμε πέρας Απορρίπτεται. 245 υπέρ. Κατά. Έλεγχος. 245. Ψηφίζουμε. Α, μισό λεπτό, λέει ο Πρόεδρος. Συμπαθάτε με. Και το 245 δεν είναι. Ναι. 2.45. Αυτό ψηφίσαμε. Και έχει εγκριθεί. Πέρασε. Πάμε τώρα στην αιτιολογική παράγραφο 5 και τροπολογία 4. Υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική B. Υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. 249 και 250 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 251 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 252 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 254 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 255, 256 και 257 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 253 καταπίπτει 258 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται, 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 259 υπέρ κατά αποχές Έλεγχος για το 259. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται με 29 ψήφους κατά. 260 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 261 υπέρ, κατά, αποχές Απορρίπτεται, νομίζω όλος κάνουμε έλεγχο το 261. Πέρασε ο φορείος. Εγκρίνεται με πέντε ψήφους διαφορά. 6 καταπίπτει. Πάμε στην συμβαστική Συ, Υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. 1967 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 7 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος για το 7. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορρίπτεται. 68 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική D υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική E υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 279 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Διακοσία υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 281 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 9. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 282 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 285 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική F. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 289. υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μια γλωσσική τροπολογία που αφορά το 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 200 91 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 14 καταπίπτει. 292 καταπίπτει. 293 καταπίπτει. Και 290 επίσης, μήπως πρέπει να την ψηφίσουμε. Αν να την ψηφίσουμε. 294 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται και τώρα ψηφίζουμε το σύνολο του σχεδίου της νομοδότης όπως τροποποιήθηκε με νομαστική ψηφοφορία ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι, πέρας. Εγκρίνεται. 46, 0, κατά. Ευχαριστούμε τον εισηγητή για τη δουλειά του. Σας ευχαριστώ που ήρθατε πέρα στις συνεδρίες. Next meetings, I'll just uh, uh remind you επόμενη συνεδριά σας υπενθυμίζω, 11 και 12 Απριλίου στις Βρυξέλλες και 25 Απριλίου πάλι στις Βρυξέλλες. Ευχαριστώ.